ε, εκθέσεις ε, της βραδιάς. Ε, συνάδελφοι, 10 λεπτά κατά μέσο όρο ανά έκθεση για να τελειώσουμε ε, στις 12. Γίνεται καταρχήν. Λοιπόν, σύντομη παρουσίαση των ακόλουθων εκθέσεων. Πρώτα απ' όλα, Σάιμον Μπουσούτιλ, κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη, αρχέ, ενέργεια και μέσα. Να δώσω το λόγο στον εισηγητή μα για τέσσερα λεπτά. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν σε δύο προτάσεις θα έπρεπε να συνοψίσω, θα έλεγα ότι η Ευρωβουλή είναι υπέρ και μάλιστα στεναρά υπέρ όλων αυτών των μέτρων για την κοινή πολιτική μετανάστευση. Δεύτερον, ότι η Ευρωβουλή δεν θέλει μια κατακαιρματισμένη πολιτική στην προσέγγιση στα θέματα μετανάστευση, αλλά μια συνεκτική, συνολική πολιτική. Αυτή η συνεκτική πολιτική μπορεί να είναι αποτελεσματική. Και τα λέω αυτό υπό το φω των πρόσφατων επίκαιρων περιπτώσεων. Αυτών που είδαμε σε σχέση με το πλοίο Πινάρ που έσωσε, 140 μετανάστες σε διεθνή ύδατα. Αυτό τι δείχνει. Αυτή η περίπτωση δείχνει ανάγλυφα πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια κοινή μεταναστευτική πολιτική, μια κοινή με άλλα λόγια πολιτική. Μας δείχνει αυτή η περίπτωση το αντίτιμο το οποίο πρέπει να πληρώσουμε στα όσα θα πρέπει να κάνουν, στα όσα συμβαίνουν, γιατί δεν έχουμε ακόμα μια κοινή μεταναστευτική πολιτική. Ο κάθε ένας απεμπολεί ευθύνε ε, τις μεταθέτει σε άλλους ε, και κάθε ένας δακτυλοδικτύος υπεύθυνου άλλους ε, χωρίς να καταλήγουμε σε μια επαρκή ικανοποιητική λύση. Ταυτόχρονα συνεχίζουν να πνίγονται και να πεθαίνουν κάθε μέρα άνθρωποι μπροστά στα μάτια μας. Πρόεδρε, είναι ντροπή, είναι έσχος αυτό που συμβαίνει. Μια χώρα 60 εκατομμυρίων να προσπαθεί να μεταθέσει τις ευθύνες ε, σε σχέση με τις διατάξεις σε μια χώρα με λιγότερο από ένα εκατομμύριο, με λιγότερο από μισό εκατομμύριο κατοίκους, ε, στη Μάλτα δηλαδή από πλευρά της Ιταλίας. Και γι' αυτό θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη αυτή την κατάσταση και πριν από τις ευρωεκλογές ε, αυτό έχει πάρα πολύ ε, έντονο οξύ χαρακτήρα. Όμως ε, δεν είναι δυνατόν ε, να κλείσουμε τα μάτια και να μην είμαστε σε υπέρ μιας θετικής προσέγγισης μια και κατέστη εφικτό να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα των μεταναστών που βρισκόντουσαν στο πλοίο Πίνα. Μια παρέμβαση, μια παρέμβαση που έγινε με βάση τον κοινό νου την λογική για τον σεβασμό των διατάξεων και να μην επιβληθεί ο νόμος της Σούγκλας. Ελπίζω λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορεί να μεταθέτει κανείς τις ευθύνες και δεν θα, μπορεί να, δεν θα πρέπει να δακτυλοδικτύωσει υπεύθυνου άλλους. Αυτό δεν εξυπηρετεί καμιά λύση. Μια κοινή πολιτική είναι η λύση που θα οδηγήσει σε διευθέτηση των πραγμάτων. Μια συνολική παρότι επώδυνη και δύσκολη λύση. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θέλω εγώ να επισύσω την προσοχή στο ότι υπάρχει αυτή η ανθρώπινη τραγωδία στην διάσταση αυτού του προβλήματος μια και πρέπει να σταματήσει εξάπαντος η παράνομη μετανάστευση. Και ο επιμερισμός βαρών όσον αφορά τα θέματα μετανάστευσης θα πρέπει άμεσα να επιτευχθεί και θα πρέπει να είναι ένα νομικά δεσμευτικό μέσο. Επίσης, τρίτον, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σπουδαιότητα στην επιστροφή ε, των παράνομων μεταναστών ε, στις χώρες τους και να υπάρξουν συμφωνίες όσον αφορά τις τρίτες, τρίτες χώρες ώστε να μπορούν να καλύπτονται τέτοιου είδους περιπτώσεις ε, παράνομων μεταναστών και η υπηρεσία Frontex θα πρέπει να ενδυναμωθεί όχι μόνο οικονομικά αλλά κυρίως όσον αφορά τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Και τέλος προσθέτω ότι θα πρέπει να εντείνουμε την μάχη των αγώνα που δίνουμε κατά του οργανωμένου εγκλήματος και καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές προτάσεις σε, διάφορα σημεία. Απομένει ένα σημείο το οποίο είχε απομείνει λόγω της πλειοψηφίας της σοσιαλιστικής ομάδας για τα, το δικαίωμα χωρίς ψήφου στους μετανάστες. Κάτι που θεώρησα ότι δεν μπορούσε να ήταν αποδεκτό για μένα και γι' αυτό υπέβαλα μια εναλλακτική λύση ώστε θα υπάρξει μετατροπή αυτού, αυτής της πρότασης σε μια συμβαστική πρόταση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Πουζούτιλ για την σημαντική του έκθεση μια έκθεση η οποία έχει ως κεντρικό θέμα την περαιτέρω ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και συγκεκριμένα την κοινή μεταναστευτική πολιτική για την Ευρώπη. Όπως αναφέρεται και στην έκθεση, το σύμφωνο για τη μετανάστευση, το οποίο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ε, ε, δίνει μια κατεύθυνση σε σχέση με την πολιτική μετανάστευση και ασύλου. Λαμβάνονται κάποιε δεσμεύσει, οι οποίε θα πρέπει τώρα να υλοποιηθούν στην πράξη. Τον επόμενο μήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει μία μέθοδο μέσω τη οποία θα είναι δυνατόν να παρακολουθείτε η υλοποίηση του συμφώνου με τίσχε εκθέσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να διαρθρωθεί η ετήσια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη μετανάστευση και τις πολιτικές ασύλου από το 2010 και μετά ο ορισμός ε, της, ε, των γενικών στόχων πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται στο σύμφωνο, θα γίνει στο πλαίσιο του επόμενου πολιετού προγράμματος, προγράμματος της Στοκχόλμης, το οποίο θα εγκριθεί φέτος επί Σουηδικής Προεδρίας. Η έκθεση Μπουσούτιλ δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ χρήσιμα στοιχεία και για τη δική της συνεισφορά που θα είναι υπομορφή ανακοίνωση που θα πρέπει να ε, μάλλον να εγκριθεί πριν από το καλοκαίρι. Με ικανοποίηση σημειώνω ότι υπάρχει εν γέννη σύγκληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται από την έκθεση Μπουσούτιλ να δράσει και πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρά σε πολλούς από τους τομείς αυτούς, παραδείγματος χάρη ε, για τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων και της ανάλυσης δεδομένων. ανάλυση των κινδύνων λαθρομετανάστευσης και συνεργασία με τρίτες χώρες, ενίσχυση της νόμιμης μετανάστευσης. Αναφέρω έναν τομέα συγκεκριμένο που ο κύριος Μπουσούτηλ εκφράζει κάποιες ανησυχίες. Αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα μετανάστευσης. Όπως αναφέρατε και εσείς κύριε Μπουσούτη στην παρέμβασή σας, πρόσφατα γεγονότα στην Μεσόγειο τόνισαν και επεσήμαναν ακόμη πιο έντονα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Πρέπει να σας ε, διαβεβαιώσω κύριε Μπουσούτηλο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι δεσμευμένη στο να βρεθεί μια λύση που θα υποστηρίζει τα κράτη-μέλη που δέχονται έντονες μεταναστευτικές πιέσεις. Ένα παράδειγμα. εν ώψη και του κανονισμού του Δουβλίνου. Ε, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και θα γίνουν οι απαραίτητε τροποποίησεις ώστε να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένη πίεση. Υπάρχει επίσης το Γραφείο Ασύλου που θα υποστηρίζει τα μέλη αυτά και θα δοθούν και κονδύλια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αύριο ε, θα γίνει το μεσημέρι ψηφοφορία και τώρα έχουμε μια σύντομη παρουσία τη έκθεση τη κυρία Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλη για τον έλεγχο τη δημοσιονομική εκτέλεση του μηχανισμού προενταξιακή βοήθεια. Κύριε Συγγετρή. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου καταρχά να επενθυμίσω ότι ο μηχανισμό προενταξιακή βοήθεια είναι ο νέο δημοσιονομικό μηχανισμό